Die Sitzung ist eröffnet. Άρχεται η Πρώτο θέμα είναι το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας. Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το πρόγραμμα.